Okay, colleagues, are people happy we start the vote? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Είναι 9 και 10. Καλώς ήρθατε. Θα ξεκινήσουμε με το 9. Δημοσιονομικοί κανόνες. Είμαι εισηγήτρια πάνω σε αυτό. Οι συζητήσεις έχουν γίνει, δεν θα πω πολλά. Εκτός από το ότι οι τροπολογίες τις οποίες ψηφίζουμε ενισχύουν τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα καταπιστεύματα, τον έλεγχό τους, το υπόλογο τους και την οργάνωσή τους. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μέσω των συμβιβαστικών προτάσεων τις, κατάλογε, τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Καταρχάς να κάνουμε ένα τεστ για την ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ελέγχουμε το σύστημα. Τέλος. Λείπουν κάποιοι, αλλά σιγά σιγά θα έρθουν. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 17 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 και 24 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές δεκτές. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 30 και 31 μαζί ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές δεκτές 32 και 33 υπέρ κατά αποχές δεκτές συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 και 36 υπέρ κατά αποχές δεκτές 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 37 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για την 37 Ψηφίζετε. ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες Δεκτή. 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 15 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 15 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για τη 16 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απερίφθη. Λοιπόν, ηλεκτρονική ψήφος για το σύνολο του ψηφίσματος. Ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας συνάδελφοι. Θα στείλουμε τη γνωμοδότησή μας αυτή στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Περνάμε στο σημείο 10 τώρα. Δημοσιοποίηση φορολογικών πληροφοριών από συγκεκριμένες επιχειρήσεις τύπους και θηγατρικές. Σλάιν, Έλλη, θες κάτι να μας πεις πριν την ψηφοφορία. Περνάμε στην ψηφοφορία λοιπόν, ξεκινάμε με την 6 υπέρ, κατά, αποχές, Α, απορρίπτεται. Ψηφίζεται ηλεκτρονικά μάλλον, ηλεκτρονική κλίση ψηφίζεται, πέρα της ψηφοφορίας, δεκτή. 48 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 50 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη. 8 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 8. Υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Ε, ψηφίζουμε. Νομίζω ότι τα μπλέξατε λέει. Πρόεδρος, ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή. Κοιτάξτε, έχουμε πολλές ψηφοφορίες, πρέπει να μπούμε στον αριθμό. Εννέα υπέρ, κατά, αποχές Δεκτή. 54 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη. 10 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 11 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 11. Ψηφίζετε παρακαλώ. Τέλος. Δεκτή. Συνάδελφοι πρέπει να φαίνεται το τι ψηφίζετε. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 58 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 59 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 60 υπέρ, α όχι, έχει καταπέσει 60, 13 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 14 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 15 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 16 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 17 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 62 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 63 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 64 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 65 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 66 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 65 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή, θεωρείται δεκτή 25. Λοιπόν 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 68 υπέρ κατά αποχές απερίφη. 69 υπέρ κατά αποχές απερίφη. 27 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 27 παρακαλώ ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 70 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 28 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 28 ψηφίζουμε τέλος απερίφθη 28 71 υπέρ κατά αποχές απερίφη 72 υπέρ κατά αποχές απερίφη 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 73 υπέρ κατά αποχές απερίφη 30 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 30 τέλος της ψηφοφορίας απερίφθη 31 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές δεκτή. 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 37 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 38 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 38 υπέρ κατά αποχές απερίφθη Τριάντα υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 40, υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 40 ψηφίζεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Δεκτή. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 4. Ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 5. Ψηφίζεται παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας απερίφθη. 46 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 47 Λοιπόν, 47 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Και τώρα ψηφίζουμε για το, το σύνολο ονομαστική κλίση ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια στην κυρία Στάιν. Έχετε το λόγο κυρία Στάιν. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συνεργασία που επέδειξαν είναι καλό η Επιτροπή μας να έχει κάποιο λόγο σε σχέση με αυτό το θέμα, γιατί οι εκθέσεις αναχώρα είναι βασικές για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Και εμείς είμαστε ε, εναντίον κάθε μορφής φοροδιαφυγής, οπότε είναι σημαντικό να έχουμε τα σωστά στοιχεία και νομίζω ότι θα πρέπει να το γνωστοποιήσουμε με την τεράστια πλειοψηφία που είχαμε σε αυτό και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περνάμε τώρα στην αυστηρότητα σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες της εξωτερικής ε, δράσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι η συγγήτρια. Έχουμε Μία ε, προφορική ερώτηση, τρει τροπολογίε από την Μαρία Χόιμπουχ. Ε, πρώτα ξεκινούμε λοιπόν με την προφορική ε, τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όλη την ερώτηση, όχι με ονομαστική, άρχεται η ψηφοφορία. Ας το κάνουμε με ονομαστική. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίες Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στο ψήφισμα. Δεν ξέρω ε, εάν επειδή ε, ούτως ή άλλως υπάρχει και μια εισηγήτρια για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, ε, παρόλο που είμαι εγώ εισηγήτρια, αν θέλει να μιλήσει, όχι. Οπότε ε, πρέπει να σα πω ότι είναι πολύ σημαντικό να εγκρίνουμε αυτή τη γνωμοδότηση για να επηρεάσουμε την Επιτροπή πριν δημοσιεύσει τη δική τη πρόταση. Η τροπολογία 29 υπέρ αποχέ απορρίπτεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Είναι χωριστή ψηφοφορία μάλλον. Μέρος πρώτο. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 36. Άρχεται η ψηφοφορία. vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε τη 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε τη 48 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε τη 49 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 53. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 σε τμήματα, πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Το πρώτο τμήμα της 55 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56. Υπέρ. Να ελέγξουμε για να δούμε το αποτέλεσμα. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 55. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Α, συγγνώμη. Σε τμήματα. Τμήμα 1. Της 60 υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Έχετε την κατάλογο με τις ψηφοφορίες. Είναι αργά. Ε, Πέρα της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. οικονομική βία έχει εξαιρεθεί, κύριε Πρέντα. Αυτό είναι το δεύτερο τμήμα στην ουσία. Εξαίρεση αυτής της φράσης. Δεύτερο τμήμα της ε, τροπολογίας 60. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Είχε απορριφθεί ούτω ή άλλω, λοιπόν, είχαν απορριφθεί οι λέξει. Οι σοσιαλιστέ και το ΕΛΚ ήταν κατά, άρα απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε την 63. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία, Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε συμβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 73 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 73 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ξαναδώ. 74 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε την 75. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πες τις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε. 76 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. 76 πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 77. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 24 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ απο, κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 28 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ήταν πολύ κοντά το αποτέλεσμα. Το ψήφισμα συνολικά με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας, συνάδελφοι, γι' αυτό. Και πάμε τώρα μια μικρή αλλαγή έχουμε τον προσωπικού έχουμε τη συμπερίληψη των εκπομπών ε, αερίων του θερμοκηπίου για την χρήση την αλλαγή χρήσης γης, ε, την ε, δασοκομεία στο πλαίσιο του 2030. Ο κύριος Μαρσελές δεν είναι εδώ, που είναι εισηγητής, άρα δεν θέλει να πει κάτι, άρα ξεκινούμε με την τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 8, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Όσοι θέλουν να ψηφίσουν την 8, πέρα στις ψηφοφορίες, απορρίπτεται. Πάμε στη 40 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Να το ξανακάνουμε, 40 υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω απορρίπτεται. Να ελέγξουμε όμως τη 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Νομίζω εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. Να σε ελέγξουμε την 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 9. Ψήφισαν όλοι Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται 39 και πάλι. Όλο το ίδιο θα είναι μου φαίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά απόχέ Να ελέγξουμε την 11. Νομίζω όμω ότι την ίδια πλειοψηφία θα έχουμε και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία Όχι, απορρίπτεται. Πρέπει να τα κάνουμε όλα χωριστά γιατί είναι πολύ κοντά τα αποτελέσματα. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε τη 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Δεν ψηφίσατε όλοι. Αν θέλετε να ψηφίσετε, ψηφίστε τώρα. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε τη 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε τη 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά. Το ίδιο. Ας ελέγξουμε την 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι διαφορετικά τώρα. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε τη 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε τη 19. Άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 19. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Την 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε τη 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία, απορρίπτεται. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. απόχέ. Ελέγχουμε την 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Είμαστε στην 3. Ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές έχουμε την 5 άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ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 τη γνωμοδότηση συνολικά με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Σας ευχαριστούμε πολύ και τον ε, ε, Φλωράν ε, Μαρσελέση. Συνάδελφοι, ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες. Αν φεύγετε, παρακαλώ φύγετε με ησυχία. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, περιμένουμε τον ε, εισηγητή. Η ψηφοφορία πήγαινε πιο γρήγορα από ό,τι είχα υπολογίσει και ο εισηγητής δεν έχει έρθει ακόμα. Θα έπρεπε να την είχα καθυστερήσει λίγο. Colleagues, our rapporteur... Συνάδελφοι, έχει καθυστερήσει ο εισηγητής, μου είπαν ότι θα έρθει στις 10 και 10. Προτείνω να διακόψουμε μέχρι τις 10 και 4. Είναι καλύτερο να πάτε για καφέ αντί να περιμένετε. Ούτε η Επιτροπή έχει έρθει. Ο εισηγητής θα έρθει στις 10 και 10 και θα ξεκινήσουμε στις 10 και 4. Το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη ούτως ή άλλως έχει διαγραφεί, διαγράφτηκε χθες, επομένως ε, διακόπτω τη συνεδρίαση μέχρι τις 10 και 4.

Συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε την εξέταση του επόμενου σημείου στην ημερήσια διάταξη παρουσία του κυρίου Γκέρενς. Ευχαριστώ για την υπομονή σας, ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Πάμε λοιπόν στο σημείο 13, Γενικός Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018. Πρόκειται για την πρώτη μας συζήτηση. Έχουμε τον Γενικό Εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είστε εδώ, κύριε Γκέρενς και κύριε Μούρεσαν. Είναι εδώ και ο κύριος Μούρεσαν. Έχουμε και το δικό μας εισηγητή, τον κύριο Σάρλο Γκέρενς, θα ακούσουμε όμως πρώτα τον κύριο Μούρεσαν που είναι γενικότερος εισηγητής για το θέμα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά τον εισηγητή της Επιτροπής μας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κανένα πρόβλημα κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε σήμερα το πρωί. Να σας μιλήσω. Και ήθελα να σας μιλήσω στην αρχή αυτής της διαδικασίας, της δημοσιονομικής, Τώρα πηγαίνω σε όλες τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συζητήσουμε γενικότερα τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ακούσω από τα μέλη των επιτροπών τι είναι το σημαντικό στο κάθε φάκελο αρμοδιοτήτων. Έτσι ώστε πρώτον να τα λάβω αυτά υπόψη μου στα επόμενα στάδια της διαδικασίας και δεύτερον να ε, βεβαιωθώ ότι όταν το Κοινοβούλιο οριστικοποιήσει τη θέση του εν ώψη των σημαντικών διαπραγματεύσεων που επίκυνται με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να είμαστε σίγουροι ότι τα πιο σημαντικά σημεία της Επιτροπής σας θα έχουν συμπεριληφθεί. Πού βρισκόμαστε λοιπόν στη διαδικασία για το προπολογισμό. Στις αρχές Φεβρουαρίου παρουσίασα το σχέδιο έκθεσης για τις κατευθυντήρες γραμμές για το προπολογισμό για το 2018 στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για τις συνολικές πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάσει το σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο θα κάνει ε, στα τέλη Μαΐου. Στην Ολομέλεια του Μαρτίου υιοθετήσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές μου και περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο προϋπολογισμού στα τέλη Μαΐου πριν εκφράσουμε τη θέση μας επ' Ποιε θα πρέπει να είναι οι πολιτικέ προτεραιότητες για τον προπολογισμό τη Ένωσης για του χρόνου, κατά την άποψή μου. Η απάντηση είναι διτή. Πρώτον, ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης και δεύτερο, ασφάλεια των πολιτών. Αυτές είναι οι πολιτικέ προτεραιότητε, αυτά περιμένουν από εμά οι πολίτε της Ευρώπη, υπαριθμόν ένα δουλειέ, υπαριθμόν δύο ασφάλεια. Άρα, πρέπει τους περιορισμένους οικονομικούς μας πόρους να τους αξιοποιήσουμε ε, για να πετύχουμε ορισμένα αποτελέσματα. Ω προ το πρώτο, ανάπτυξη και θέσεις απασχόληση. Νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε τα πιο αξιοσημείωτα αποτελέσματα ενισχύοντα την οικονομία τη Ένωση, καθιστώντα την πιο αποτελεσματική, ενισχύοντα την έρευνα, την κοινοτομία, την καινοτομία της μικρομεσαίας επιχειρήσεις, τι υποδομέ, ενισχύοντα τον ορίζοντα 2020, τα προγράμματα διασύνδεοντας την Ευρώπη, Connecting Europe Facility, το πρόγραμμα COSME και διάφορα άλλα προγράμματα προγράμματα για τη μείωση της ανεργίας των νέων. Και κάτι που αφορά περισσότερο εσάς, ε, ασφάλεια των πολιτών. Ε, δύο συναισθώσεις. Πρώτον, ε, δύο α αν θέλετε εσωτερική ασφάλεια, δύο β εξωτερική ασφάλεια, γιατί δύο α εσωτερική ασφάλεια πρέπει να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες της Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Έχουμε εργαλεία, αυτό που διαθέτουμε είναι οι διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αξιοποιούν τους περιορισμένους μας πόρους και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα με τα κονδύλια. Να ενισχύσουμε τις διάφορες υπηρεσίες και γραφεία της Ένωσης, να στηρίξουμε τα πιλωτικά προγράμματα στον τομέα της αμήνης, έτσι όπως θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και δύο β εξωτερική ασφάλεια πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή στο άμεσο γειτονικό μας περιβάλλον. Γιατί από εκεί εκπορεύονται κατά βάση οι προκλήσεις. Μιλούμε για την ανατολική γειτονία, έχουμε μια πιο, όλο και πιο ενεργή Ρωσική Ομοσπονδία, Ρωσική Ομοσπονδία όλο και πιο ενεργή και προς τον Νότο πρέπει να στραφούμε στην άμεση γειτονιά μας, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των μεταναστών με τις προσφυγικές ροές που βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια. Και η δράση μας πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη των στόχων για την αηφόρο ανάπτυξη ε, βάσει της πολιτικής ατζέντα για το 2030 και πρέπει φυσικά να αναγνωρίσουμε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια είναι εξίσου σημαντική τουλάχιστον, γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι κατά βάση οι μεγαλύτεροι δωρητές. Είμαστε μακριά από το 0,7% του GNI που δεσμευτήκαμε να συμβάλλουμε, ωστόσο οι πρόσφατες εξελίξεις είναι θετικές και γι' αυτό Στόχος μας είναι να έχουμε επαρκή χρηματοδότηση για την ανθρωπιστική βοήθεια και για τις αναπτυξιακές δράσεις, να μπουν αυτά στο προϋπολογισμό του 2018. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας. Αυτό είναι το σημαντικό, με τους υφιστάμενους πόρους πάντοτε. Υπ' αυτή την έννοια, στις 11 σήμερα το πρωί στην Επιτροπή για τον Προϋπολογισμό θα συνεδριάσει η ομάδα εποπτείας των μέσων και εργαλείων εξωτερικής χρηματοδότησης η οποία θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα με τους υφιστάμενους πόρους. Έχουμε το EFSD, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αϊφόρο Ανάπτυξη, είναι ένα εργαλείο εξαιρετικά σημαντικό που μπορεί να καλύψει κάποιες από τις ελλείψεις στην οικονομική βοήθεια ο προϋπολογισμός θα συμβάλλει κατά 350 εκατομμύρια ευρώ ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την αηφόρο ανάπτυξη και στον τριμερή διάλογο το περασμένο φθινόπωρο. Είπαμε ότι θα ενσωματώσουμε τα ποσά αυτά στο προπολογισμό αρχή γενομένη του 2017, άπαξ και αποκτήσουμε τη νομική βάση. Και όπω γνωρίζετε, κυρία Πρόεδρε, εσεί προεδρεύσατε χθε στη συνεδρίαση τη διευρυμένη Επιτροπών ΑΦΕΤ Εξωτερικών Υποθέσεων και ε, Προπολογισμού. Εγκρίναμε λοιπόν την έκθεση. Μόλις υπάρξει λοιπόν η νομική βάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει σχέδιο τροποποίησης του προϋπολογισμού που θα κινητοποιήσει τα κονδύλια που έχουν κατανεμηθεί για το 2017 Μιλούμε για 275 εκατομμύρια που έχει προβλεφθεί να κινητοποιηθούν πάνω από την οροφή του ε, τίτλου 4 και θα πρέπει να πράξουμε και τα δέοντα αντίστοιχα για το 2018. Περιμένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει τα ποσά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αεφόρο Ανάπτυξη στο σχέδιο προϋπολογισμού που θα παρουσιάσει στα τέλη Μαΐου και εάν η νομική βάση εγκριθεί εγκαίρως, τότε θα είμαστε σε θέση να εγκρίνουμε το σχέδιο προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη διαδικασία συνδιαλλαγής το φθινόπωρο του 2017. Κάτι που δεν μπορέσαμε να πράξουμε πέρσι το φθινόπωρο γιατί υπήρχαν καθυστερήσεις λόγω απουσίας νομικής βάσης. Τώρα θα έχουμε σχέδιο τροποποιητικό του προϋπολογισμού και θα καταστούν όλα αυτά εφικτά. Η αναθεώρηση του ε, πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, η ενδιάμεση αναθεώρηση ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή και σύμφωνα με αυτήν έχουμε άλλα 20 εκατομμύρια ε, ευρώ στο αποθεματικό για έκτακτες καταστάσεις. Από τα 280 εκατομμύρια ευρώ πήγε αυτό το αποθεματικό στα 300 και αυτό είναι καλά νέα. Και καταλήγοντας τις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις θα ήθελα να μιλήσω εν συντομία για τα καταπιστεύματα, trust funds. Ε, στην Επιτροπή Προϋπολογισμού εξ αρχής ε, εντοπίσαμε την ανάγκη ε, δημιουργίας αυτών των καταπιστευμάτων. Βεβαίως μας ανησυχεί, δεν θέλουμε ο προϋπολογισμός να χάσει την ολότητά του, τον ενιαίο του χαρακτήρα, την ενότητά του, όμως πρέπει να διασφαλιστούν και τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Μας ενδιαφέρουν οι υποσχέσεις, pledges. Εμείς έχουμε υποσχεθεί 1,8 δις ευρώ στο καταπίστευμα mandat και 117 εκατομμύρια ευρώ είναι μια κατάσταση μη βιώσιμη, είναι θέμα αξιοπιστίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολιτικές υποσχέσεις των κρατών μελών, ε, δεσμεύσεις ε, να εκπληρώνονται. Και από πλευράς Επιτροπής Προϋπολογισμού πέρσι το Μάιο ασχοληθήκαμε με την Ιορδανία και το Λίβανο. Είδαμε ότι οι πόροι βάσει της έκθεσης ε, έχουν ήδη πάει επιτόπου και βοηθούν στο τομέα της εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, στην εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό η προβλεψιμότητα. Θα πρέπει όσοι, ε, όσοι δουλεύουν επί τόπου να έχουν προβλεψιμότητα. Το Μάιο να γνωρίζουν αν θα τους έρθουν οι πόροι την επόμενη χρονιά για να μπορέσουν να ξαναπροσλάβουν καθηγητές και να υπάρχει συνέχεια στο εκπαιδευτικό, στο διδακτικό έργο. Άρα μας ενδιαφέρει να είμαστε ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται και αξιοποιούνται όλα αυτά τα καταπιστεύματα. Ο αρμόδιος επίτροπος απέστειλε επιστολή στη σχετική επιτροπή καλώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλακεί, να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων, των διοικητικών ομάδων, αν θέλετε steering boards, των ομάδων που δίνουν τις κατευθύνσεις σε αυτά τα καταπιστεύματα για να διατηρηθεί και να διασφαλιστεί η συνέχεια και από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή η πόρτα είναι ανοιχτή, μας έχουν ανοίξει την πόρτα να πάμε να συμμετάσχουμε και θα πρέπει να το πάρουμε το θέμα στα σοβαρά. Και τέλος κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να αναφερθώ στα πιλωτικά προγράμματα. Εγώ επιθυμώ να χρηματοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο το δυνατόν περισσότερα πιλωτικά προγράμματα και όσο το δυνατόν περισσότερο. Και πώς θα το επιτύχουμε αυτό. Με τον εξή τρόπο θα εξετάσουμε μόνο τα πιλωτικά προγράμματα που έχουν σταλεί για προαξιολόγηση, για έγκαιρη αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όποιο θέλει να προχωρήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα, Επιτροπή, όποιο και αν είναι αυτό, κοινοβουλευτική ή οποιοδήποτε άλλο φορέα, πρέπει να το στείλει στην Κομισιόν για pre-assessment, εκ των προτέρων για πρώτερη αξιολόγηση. Και καταληκτική προθεσμία είναι η 3η Μαΐου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα τα σημειώσει αυτά τα πιλωτικά προγράμματα που έχει δεχθεί και έχει λάβει για εκ των προτέρων αξιολόγηση και λαμβάνοντας υπόψη τι υποβάλλετε εσείς ως προτάσεις και σε συνεργασία με όλες τις πολιτικές ομάδες και όλους τους εισηγητές στην Επιτροπή Προϋπολογισμού θα φτιάξουμε ένα καλάθι πιλωτικών προγραμμάτων που θα είναι επιλέξιμα προς στήριξη. Είναι πιο εύκολο για εμάς να δουλέψουμε αν μας προτείνετε λίγα όμως εγώ θέλω να μας προτείνετε πολλά για να κάνουμε και εμείς όσο το περισσότερα και να καλύψουμε όσο το περισσότερα. Άρα σας καλώ να μας υποβάλλετε πολλές προτάσεις για πολλά πιλωτικά προγράμματα, αλλά να μην ξεχάσετε να τα στείλετε και στην Κομισιόν για εκ των προτέρων αξιολόγηση, γιατί μόνο αυτά που θα έχουν περάσει από την Κομισιόν έχουν πιθανότητες να τύχουν έγκριση από εμάς στη συνέχεια. Αν λάβετε το καλό βαθμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, α ή β, πάρετε είναι πολύ ψηλέ οι πιθανότητε. η πρότασή σας να συμπεριληφθεί στο τελικό καλάθι, στο... Ε, στη συνολική δέσμη των πιλωτικών προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν και θα στηριχθούν. Άρα, από τη δική σας Επιτροπή περιμένω να λάβω προτάσεις για ενδιαφέροντα πιλωτικά προγράμματα και δράσεις. Και επαναλαμβάνω, καταληκτική προθεσμία είναι η 3η Μαΐου για να τα στείλετε για εκ των προτέρων αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά, κυρία Πρόεδρε, είχα να πω. Ε, περιμένω στενή συνεργασία και αλληλεπίδραση με όλους εσάς μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Σήμερα είναι η αρχή της ε, ε, συνεργασίας μας και της επικοινωνίας μας. Επαναλαμβάνω με δύο λόγια αυτό που νομίζω ότι ενδιαφέρει όλους είναι οι δουλειές, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η ασφάλεια των πολιτών. Είμαι εδώ κατά κύριο λόγο για να σας ακούσω και περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω τις απόψεις και τις προτάσεις σας. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ για την πολύ σαφή παρουσίαση των προτεραιοτήτων σας. Σήμερα το πρωί ψηφίσαμε για τον οικονομικό κανονισμό, για τα καταπιστεύματα. Νομίζω ότι για πολλά θέματα ε, συντασσόμαστε και συμπορευόμαστε. Έχουμε όμως τον Σάρλ Γκέρενς που είναι εισηγητής για την Επιτροπή μας. Παρακαλώ. Να ευχαριστήσω τον Γενικό Εισηγητή που έθεσε το δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε έναν ρόλο τομεακό εμείς να παίξουμε και χαίρομαι που έχουμε τον Γενικό Εισηγητή μαζί μας για να ακούσει τις δικές μας επιθυμίες. Ο προϋπολογισμός είναι ένα πολιτικό μέσο, μεταφράζει με αριθμητικό τρόπο στην πραγματικότητα τις πολιτικές προτεραιότητες, τις υποχρεώσεις, τις πολιτικές που έχουν αναλυφθεί εφόσον υπάρχουν και οι οποίες καλούνται μέσω των δημοσιονομικών ρυθμίσεων να γίνουν αξιόπιστες ή όχι. Δεύτερη παρατήρηση, θα πρέπει να δούμε τον προϋπολογισμό με βάση τους πολιτικούς του προσανατολισμούς, προσανατολισμούς τους οποίους έχουμε αποφασίσει στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμίζω εδώ, θέλει να παραμείνει η πρώτη δύναμη ειρήνη στον κόσμο. Υπερηφανεύεται ότι είναι η πρώτη δωρήτρια χώρα αυτό όμως θα πρέπει να συνεχιστεί γιατί από ό,τι φαίνεται μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου ε, θα, δεν θα υπάρχουν σημαντικές συνεισφορές πλέον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον προϋπολογισμό της και μάλιστα και σε εθνικό επίπεδο νομίζω ότι η αναχώρηση των Βρετανών θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα μείωσης των επιμέρους προϋπολογισμών. Θα πρέπει να δούμε επίσης τον προϋπολογισμό στα πλαίσια της πολλαπλότητα των χρηστών. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας υποχρεώνει να ασκήσουμε μια συνεκτική πολιτική και μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο, για να είναι πραγματικά συνεκτική η πολιτική αυτή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλους τους εμπλεκομένους εμπλεκομένου σε επίπεδο λοιπόν δημοσιονομικό, οι οποίοι είναι όπως είπα πολλαπλοί. Κατάρχά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της Ένωσης, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το οποίο είναι διακυβερνητικό μέσο, ανήκει σε 28 χώρες, δίδει τις πιστώσεις ε, ε, ε, του Ταμείου αυτού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό δίνει την ψευδέστηση ενός πλαισίου δημοσιονομικού ενιαίου, αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο και λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν υπηρεσία ανάπτυξης. Αλλά θα μπορούσαν να υπάρξουν και άλλοι κοινοτικοί οργανισμοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο, εθνικοί. Και από την άλλη υπάρχουν και 28 εθνικοί προϋπολογισμοί. Και να προσθέσουμε σε αυτό και τις αναπτυξιακές οργανώσεις, οι οποίες και αυτές έχουν κάποιες γραμμές που ακολουθούν που δεν είναι πάντα ευθυγραμμισμένες με τις αντίστοιχες των κυβερνήσεών τους. Πάρα πολλές φορές οι κυβερνήσεις και τα αρμόδια Υπουργεία για την Ανάπτυξη θα έλεγα συνιστούν το πολιτικό πλαίσιο αναφοράς ε, της, ε, των υπηρεσιών αυτών των αναπτυξιακών. Θα πρέπει λοιπόν οι προϋπολογισμοί να εξυπηρετούν τις βασικές μας προτεραιότητες, θα πρέπει να ψηφίζονται ε, συγκεκριμένες ε, πιστώσεις στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού και το ελάχιστο περιθώριο το οποίο παραμένει θα πρέπει φυσικά να το ε, διεκδικούμε. Πόσο μάλλον που εάν πράγματι θέλουμε να παίξουμε ρόλο σε επίπεδο πολιτικό, θα πρέπει να ξεφύγουμε από το πλαίσιο αυτό έτσι ώστε όλοι να καταλήγουμε στους ίδιους στόχους. Αν κατάλαβα καλά, Υπάρχει μία αναπτυξιακή πολιτική, έτσι λέει η συνθήκη, και όχι 28 ή 30. Να προσθέσουμε εδώ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που είναι διακυβερνητικός οργανισμός και σε αυτό το επίπεδο ε, εφόσον ε, εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπάρξει μείωση του προϋπολογισμού. Το θέμα είναι αν τυχόν παραμείνει μέλος ε, στην τράπεζα αυτή. Τώρα για τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό είναι ο προτελευταίος μιας Ευρώπης 28 χωρών. Οι υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει και οι υποχρεώσεις τις οποίες οι χώρες εταίροι αναμένουν από πλευράς μας θα πρέπει, θα έλεγα, να πραγματοθούν με 27 πλέον χώρες μετά την έξοδο των Βρετανών. Θα συμφωνήσω εδώ λοιπόν με τον Γενικό Εισηγητή ότι θα πρέπει φυσικά να χαιρετήσουμε την αύξηση των 28 εκατομμυρίων που προτείνει για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω εδώ ότι αυτά κύριε Ισηγητά είναι ψίχουλα. Ψίχουλα σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες χρηματοδότησης των τροφιμικών κρίσεων στον κόσμο και της ε, ε, διατροφικής βοήθειας. Έχουμε να κάνουμε με πέντε χώρες οι οποίες ε, κατατρέχονται από ε, σειράξεις, οι πληθυσμοί τους απειλούνται από λοιμούς και δεν ξέρουμε πώς θα βγούμε από το αδιέξοδο αυτό εάν ε, η διεθνής κοινότητα και στο εσωτερικό της η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρει περισσότερα χρήματα. Και δυστυχώς παρακολουθούμε με πάρα πολλή αδυναμία ότι η κατάσταση χειροτερεύει χωρίς εμείς φυσικά να είμαστε σε θέση να δώσουμε μια δημοσιονομική ανταπόκριση. Αυτό είναι σοβαρότατο και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Είχα ξεχάσει να αναφέρω ότι ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι ο πρώτος του δεύτερου τμήματος του πολιετούς δημοσιονομικού και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, όπως να λάβουμε υπόψη επίσης και τα συμπεράσματα της αξιολόγησης της, του πρώτου τμήματος της δημοσιονομικής περίοδου μέσω της ενδιάμεσης ε, αναθεώρησης. Ένα άλλο θέμα, στο οποίο έχω αμφιβολίες για την ύπαρξη των κατάλληλων μέτρων, είναι αν θέλετε η διάχυση του προϋπολογισμού η διάχυση του προϋπολογισμού σε πάρα πολλά μικρότερα τμήματα. Απειλείται λοιπόν από διάφορους τομείς οι οποίοι δεν έχουν άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης όπως οι κλιματολογικές συνέπειες. θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα λαχείο. Η αναπτυξιακή βοήθεια έχει μια ακεραιότητα και θα πρέπει να είμαστε αυστηροί στο τι είναι η συνεργασία για την ανάπτυξη. Δεν είναι τα πάντα και με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά είναι η εκρίζωση της φτώχειας υπέρ της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το υπενθυμίζουμε αυτό από χρόνο σε χρόνο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε αυστηροί και να εφαρμόζουμε την μέθοδο QE όπως λέγουν οι Γάλλοι, δηλαδή η επανάληψη είναι η μύτη της μάθησης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν θα πρέπει λοιπόν σε καμία περίπτωση εμείς να υπαναχωρήσουμε και να αποδεχθούμε τους, να διατρέχει κινδύνους η βοήθεια για την ανάπτυξη. Απ' την άλλη να μην ξεχάσω την, τον αστερισμό θα έλεγα των ειδικών ταμείων που καθιστά ανίκανο τον παρατηρητή να έχει μια ενιαία αντίληψη για το από τι αποτελείται η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ταμεία αυτά, τα καταπιστεύματα μπορεί να χρηματοδοτούνται είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είτε από τα κράτη-μέλη, είτε από τις Εθνικές Αναπτυξιακές Υπηρεσίες, είτε από το Ταμείο για την Ανάπτυξη. Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Εγώ άκουσα να εκθέτουν τις πολιτικές τους προτεραιότητες ε, και δεν θα διαφωνήσω με αυτά, αλλά υπάρχει σαφώς ένα πρόβλημα κοινοβουλευτικού ελέγχου και φοβάμαι ότι σιγά σιγά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμερίζεται και θα εγκαταλείψει το πεδίο αυτό. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε από κοινού τους τρόπους να βρούμε μια κάποια λύση. Δεν πρέπει να αγνοούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Πρέπει να δείξουμε ότι κατανοούμε το πρόβλημα και δεν θα αφήσουμε να μας επιβάλλουν τέτοιου είδους καταστάσεις. Θα πρέπει να μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περισσότερη διαφάνεια, για περισσότερη προβλεψιμότητα, γιατί ο προϋπολογισμός δεν είναι κάτι το γενικόλογο και το θολό. Είναι συγκεκριμένο, όχι μόνο σε σχέση με τους αριθμούς, αλλά και σε σχέση με τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Τώρα, ε, το τι θα ήθελα να πω σε σχέση με το σεβασμό των υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει. Είναι σαφές ότι αν δεν μπορέσουμε εμείς εδώ να πείσουμε και να καλέσουμε τους εκπροσώπους των 28 χωρών να μας πούν τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να πετύχουν τους στόχους, στους οποίους θυμίζω έχουν συμφωνήσει, έχουν δεσμευτεί, έχουν δώσει εντολή στους διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάνε στο Άντις και να πούνε το ποια θα είναι η πολιτική μας. Και μετά δεν κάνουν τίποτα και δεν δίνουν τίποτα, μας δουλεύουν κοινώς. Οπότε θα πρέπει να μην χάσουμε την αξιοπιστία την οποία έχουμε, έστω και κατελάχιστον. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να έχει μία άποψη με ξεκάθαρο τρόπο. Αυτές είναι οι απόψεις που έχω. Εύχομαι καλή δουλειά στον συνάδελφο και ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την διαδικασία. Ε, θυμούμε τον κύριο Αρτουή που μου είχε δώσει ένα πρόγραμμα όλων αυτών των εξωτερικών καταπιστευμάτων και ταμείων ήταν πραγματικά ε, υπόδειγμα σύγχυσης αυτή η διασπόρα. Κοιτάξτε όλα αυτά σε σχέση με τον γαλαξία δεν σημαίνουν τίποτα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Τρεις ομιλητές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος, ε, γιατί ο Σαλ Γκέρενς ήδη είπε πολλά ουσιαστικά πράγματα για την Επιτροπή μας. Υπάρχουν όμως τέσσερα σημεία στα οποία θέλω να επανέλθω και να τον υποστήριξω και τα οποία είναι μεγάλη σημασία για εμάς. Το πρώτο είναι ότι με κάθε τίμημα πρέπει τα κράτη-μέλη να κατανοήσουν, το Συμβούλιο δηλαδή, ε, να ε, συνειδητοποιήσει την δέσμευση για το 0,7% για το 20% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Ε, είναι από το 2005 αυτό, αυτή η δέσμευση. Το 2015 έπρεπε να ε, εκπληρωθεί, δεν έγινε. Τώρα έχουμε το 2030 ε, και χρειάζεται αυτός ο δικός χάρτης για να μπορέσουμε με αριθμητικό τρόπο να δούμε πως ε, δεν θα έχουμε ένα απλό που θα μείνει στα χαρτιά, αλλά θα έχει κάποια τύχη και δεν θα έχουμε πρόβλημα και εμείς με τις αρμοδιότητές μας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, που το είπε και ο Γκέρενς, είναι ο σκοπός. Να ε, κρυζώσουμε τη φτώχεια. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία τάση που την κατανοούμε μεν, αλλά ε, υπάρχουν τόσα προβλήματα ούτως ή άλλως και χρειάζεται να βρούμε τους πόρους για όλα αυτά. Όμως αυτό που φαίνεται να γίνεται είναι ότι αυτά που προορίζονται για τη φτώχεια και την εκρίζωσή της πηγαίνουν σε άλλους ε, στόχους όπως η αηφόρος ανάπτυξη. Ε, γιατί να μην το κάνουμε αυτό μέσα από τον προϋπολογισμό της μάχης κατά της φτώχειας ή και με τη μετανάστευση και την ασφάλεια που είναι ουσιαστικά και μείζωνα προβλήματα. Δεν μπορούμε λοιπόν να μειώσουμε τα κονδύλια για την ε, εκρίζωση της φτώχειας. Θα φτάσουμε σε καταστροφικές ε, καταστάσεις όπως είπε ο Ε, Πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε πιστοί στην πολιτική μας ατζέντα και να έχουμε τις ε, πολιτικές επιπτώσεις που είναι ουσιαστικές. Να επανέλθουμε λοιπόν στον ορισμό των στόχων μας και να τους επαναδιατυπώσουμε. Τρίτον, πρέπει να λάβουμε θέση, υπόθηκε ήδη, Συλλογικά εργαστήκαμε για αυτό το θέμα, για τις επιπτώσεις του Brexit. Πρέπει λοιπόν τα ζητήματα αυτά να ληφθούν υπόψη, γιατί υπάρχουν ε, πολλές επιπτώσεις και ε, όσον αφορά στη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ηγέτη στην ανάπτυξη και στις προτεραιότητες των πολιτικών του των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέταρτον, το είπατε και πριν, είναι το θέμα των καταπιστευμάτων και του δημοκρατικού ελέγχου του Κοινοβουλίου. Είναι αυτονόητο ότι μπορούμε να ε, δούμε κατά πόσο είναι νόμιμα όλα αυτά τα καταπιστεύματα, όμως ε, θα ε, το ελάχιστο που ζητούμε συνεχώς αυτή την Επιτροπή είναι να μπουν στον προϋπολογισμό για να υπάρχει ένας δημοσιονομικός έλεγχος αυτών και να μπορεί το Κοινοβούλιο να παίξει τον ρόλο του ως ένας από τους δύο ελεγκτές του προϋπολογισμού. Αυτά τα τονίζω στην ομάδα μας και επίσης υποστηρίζω και τη θέση του εισηγητή μας σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ η Χάιντι Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Γενικό Εισηγητή. Είναι εξαιρετικό που μπορούμε τώρα να συζητήσουμε τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και τις οποίες συζητούσε η Επιτροπή εδώ και ένα χρόνο. Να πω ότι το βασικό για μένα είναι να διασφαλίσουμε ότι ο προϋπολογισμός όντως κατευθύνεται σύμφωνα με τη νομική βάση της συνθήκης της Λισαβόνας προς την εκρίζωση της φτώχειας. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι πολλά από τα χρηματιδοτικά μέσα και από τις νέες ε, προτάσεις να ε, επανακατευθύνουν τα κονδύλια προς άλλους στόχους όπως την ε, πάυση της μετανάστευσης και στην ουσία οδηγούν σε μια λανθασμένη άποψη του πλέγματος της ασφάλειας και της προστασίας. Νομίζω λοιπόν ότι αν θέλουμε να μειώσουμε ε, τις, ε, τα κονδύλια της ε, κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας μπορούμε ίσως να βοηθήσουμε τις χώρες τις αναπτυσσόμενες μέσα από τον αναπτυξιακό προϋπολογισμό και μέσα από τη συνθήκη, του στόχους που θέτει για την αναπτυξιακή πολιτική. Νομίζω ότι όντως υπήρξε αυτή η πρόοδος από το 0,7, προς το 0,7%. Όμως μια νέα μελέτη από την Κομισιόν έδειξε ότι το 1 πέμπτο της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, νομίζω αφορούσε το 2015, ε, είχε να κάνει με μετανασταυτικές δαπάνες, ε, όχι στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά σε εμάς. Δεν πρέπει λοιπόν να είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι για την πρόοδο. Και όπως είπε και ο κύριος ε, Γκέρινς πολύ καλά για τα καταπιστεύματα, θα πρέπει το Κοινοβούλιο να επιμείνει στην άποψη ότι χρειαζόμαστε μια συνεκτική ε, και έναν συνεκτικό και ενιαίο προϋπολογισμό για να πατάξουμε την φτώχεια. Σήμερα το πρωί η Επιτροπή μας ενέκρινε κάποιες ε, ενδιαφέρουσες απόψεις για τα καταπιστεύματα. Καλό τον Γενικό Εισηγητή να τα δει, διότι ε, στοχεύουν σε περισσότερους όρους ως προς την χρήση των καταπιστευμάτων για να διασφαλίσουμε αυτή την συνεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Ο Γενικός συζητητής επίσης μίλησε για την άμεση γειτονία μας. Ναι, θεωρώ ότι η εταιρική σχέση, η ανατολική εταιρική σχέση πάντοτε είχε λιγότερους πόρους από ό,τι έπρεπε, όμως δεν μπορούμε να αφήσουμε σε μειονεκτική θέση τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ε, για να ευνοήσουμε την ανατολική γειτονία, την ανατολική εταιρική σχέση. Συμφωνώ με τον κύριο Γκέρενς ότι αυτή η προσθήκη των 28 εκατομμυρίων ευρώ στην ανθρωπιστική βοήθεια είναι πολύ μικρή σε σχέση με την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχει αύξηση των διαφόρων σειράξεων που οδηγούν σε πολύ σοβαρές ανθρωπιστικές κρίσεις. Συμπεριλαμβανομένου του λοιμού που έχουμε αυτή την εποχή στην Ανατολική Αφρική, στο Σουδάν και τις υπόλοιπες χώρες. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε να, για να διασφαλίσουμε ότι θα επανέλθουμε στην τροχιά της αναπτυξιακής πολιτικής. Όπως είπε ο κύριος Γκέρενς, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει τη βασική δύναμη της ειρήνης και της ανάπτυξης στον κόσμο. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που ε, έρχονται στο προσκήνιο όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, εις βάρος των πιο φτωχών του κόσμου. Οι βίες αποφάσεις της ε, κυβέρνησης του Τραμπ που κόβουν την βοήθεια, την ενίσχυση προς τις πιο ε, φτωχές γυναίκες και παιδιά του κόσμου, μεώνοντας τα κονδύλια για την αναπαραγωγική υγεία ε, και για τα Ηνωμένα Έθνη μας οδηγούν σε αυτό. Ευχαριστώ. Στην Ιεμένη 2,2 δολάρια προορίζονταν σύμφωνα με ένα άρθρο του BBC για την τεράστια ανθρωπιστική κρίση και δυστυχώς όχι πια. Θα μιλήσουμε για τις οικογένειες σήμερα το απόγευμα και για το τι φοβερά πράγματα συμβαίνουν στην Αφρική στις 3. Ο επόμενος ομιλητής παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς ο κύριος Ρούμπικ δεν μπορεί να παραστεί στη συνεδρίασή μας και θα ήθελα να τον εκπροσωπήσω θεωρεί ότι η χρηματοδότηση αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των αναπτυξιακών ε, στόχων, των στόχων για την ανάπτυξη και πρέπει να αυξηθεί το ODA και ο στόχος του 0,7% μέχρι το 2030. Πρέπει να έχουμε στενή συνεργασία και αποτελεσματική με τον ιδιωτικό τομέα, με τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικογενειακές επιχειρήσεις και έτσι μπορεί να γίνει μόχλευση νέων πόρων για ανάπτυξη και συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και έτσι τελικά θα αυξηθεί η χρηματοδότηση που θα είναι διαθέσιμη για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μεταστείτε, μπορούμε να έχουμε ε, αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης και ενίσχυση των χωρών αυτών και να βρούμε καινοτόμους ε, τρόπους στήριξης. Ευχαριστώ, επόμενος ομιλητής, παρακαλώ. Κύριε Ισηγητά, σας ευχαριστώ για ε, τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις και για το ότι ήρθατε να μας δείτε από την αρχή της διαδικασίας για να καθορίσουμε κάποιες κοινέ γραμμές Μιλήσατε για τους ε, στόχους για την αηφόρο ανάπτυξη. Τους έχουμε συμφωνήσει με διάφορους ε, επιτρόπους, αλλά δεν μας έχει παρουσιάσει κανείς σχέδιο. Εδώ και χρόνια μιλούμε γι' αυτό. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα και να εκφραστούμε πιο επισταμένος ε, για τους στόχους αυτούς. Θα ήθελα στο σχέδιο προϋπολογισμού να είναι πιο ορατή η στόχη για την αηφόρο ανάπτυξη, με πιο ξεκάθαρες λέξεις και με πιο μεγάλη συνοχή, με στόχη με συνέπεια να αναφέρονται και με περισσότερη σαφήνεια. Θα ήθελα στο σχέδιο προϋπολογισμού να προβλεφθεί εξήγηση θα μπορούσαμε σε κάθε τίτλο να έχουμε μια μικρή διατύπωση και να λέμε ότι το συγκεκριμένο κονδύλι βρίσκεται εκεί γιατί συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων αεφόρων ανάπτυξη των SDG. Πολύ συχνά δεν κάνουμε σωστή επικοινωνία. Δηλαδή πάρα πολλοί στόχοι είναι για την αηφόρο ανάπτυξη αλλά δεν το επικοινωνούμε σωστά στον κόσμο και στην κοινή γνώμη. Συμφωνούμε με την αύξηση του 0,7% και θέλω και εγώ να συμφωνήσω με τους προηγούμενους συναδέλφους. Έχει γίνει συζήτηση για τη σταθερότητα, για την ειρήνη, για τα σχετικά καταπιστεύματα. Όλα αυτά τα εργαλεία πρέπει να χρηματοδοτούνται από διαφορετική γραμμή του προϋπολογισμού. Το έχω πει και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και να μην υφίστανται πίεση τα κονδύλια ε, της αναπτυξιακής βοήθειας. Νέες γραμμές του προϋπολογισμού ε, προβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έρευνα, για παράδειγμα. Και περικόπτεται συνεχώς ο προπολογισμό που είναι διαθέσιμος για την αναπτυξιακή βοήθεια. Όλα αυτά τα θέματα θα τα δείξουμε και στο μέλλον όταν συζητήσουμε την έκθεση. Ευχαριστώ να ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ να μιλήσει πρώτη γιατί πρέπει ο εκπρόσωπος να αποχωρήσει και μετά η άλλη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Χανιγκάλη, η Πανιγκάλη προφέρω σωστά το όνομά σας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω και πολλά να πω. Ο προπολογισμό για το 2018 δεν έχει ακόμα εγκριθεί από το Σώμα των Επιτρόπων. Θα ήθελα ωστόσο να κάνω κάποια σχόλια προκατακτικά. Πρώτον, να ευχαριστήσω θερμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ΝΤΕΒΕ για τη συνεχή αμέριστη στήριξη την οποία μας έχει προσφέρει στο παρελθόν και κυρίως κατά τη, διάρκεια, κατά τη διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού την περασμένη χρονιά. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΝΤΕΒΕ συνεχώς ασκούσε πίεση για αύξηση του προϋπολογισμού για ανθρωπιστική βοήθεια που τελικά βέβαια αυτό δεν έγινε ε, στο ε, στο τελικό κείμενο, ωστόσο ήταν πολύ θετικές εξελίξεις και ε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να μειώσουμε το βεληνικέ το μέγεθο τη κρίση στη Συρία και να αποφύγουμε το ενδεχόμενο αυτή η κρίση να εξαπλωθεί και σε γειτονικέ χώρες. Και όλα αυτά χρειάζονται στήριξη και κονδύλια. Ε, το καταφέραμε νομίζω χάρη στη στήριξη της κοινοβουλευτική Επιτροπής ΔΕΒΕ και ευχόμαστε, ελπίζουμε και περιμένουμε ότι και φέτος ε, θα ταχθούμε στο ίδιο στρατόπεδο με εσάς. Ε, αναφέρθηκε το θέμα της ενδιάμεσης αναθεώρησης και αξιολόγησης και υπήρξε συμφωνία αύξησης του προϋπολογισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυξήθηκε κατά 20 εκατομμύρια ευρώ το διαθέσιμο ποσό στο αποθεματικό για τις επίκουσες καταστάσεις για τα έκτακτα από 280 εκατομμύρια στα 300 εκατομμύρια. Άρα δεν αποτελεί αυτό μέρος του προϋπολογισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά είναι ένα συρτάρι που μπορούμε να ανοίξουμε και να βρούμε χρήσιμα εργαλεία όταν αυτό μας χρειαστεί και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτή την παρατήρηση θα ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ. Η Γενική Διεύθυνση ΔΕΠΚΟ, ο κύριος Άικ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις διαφορετικές παρεμβάσεις. Θα συμφωνήσω με όσα είπατε για την ΤΕΦΚΟ. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το οποίο έχει σημασία για τον προϋπολογισμό ο οποίος κατατέθηκε για το 2018 είναι ότι είναι συμβατός με αυτά τα οποία προβλέπονται στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε ελάχιστα περιθώρια, ενώ από την άλλη υπάρχουν συμπληρωματικά αιτήματα τα οποία φτάνουν σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό εμείς υπολογίζουμε στην δική σας υποστήριξη έτσι ώστε να υπερασπιστούμε τον προϋπολογισμό αυτό απέναντι σε όλα τα συμπληρωματικά αιτήματα τα οποία μας φτάνουν, ε, ιδιαίτερα σε σχέση και με τα SDG, θα πρέπει οι προτεραιότητες να γίνουν σεβαστές. Πολλοί από εσά αναφερθήκατε στο Brexit και στις συνέπειες αυτού. Πράγματι, νομίζω ότι ε, έχουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα πλήρη προϋπολογισμό αλλά όχι επειδή η Βρετανία θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αιτήματα δεν θα μειωθούν ε, σε σχέση με τα διαφορετικά ταμεία, ίσως να υπάρξουν κάπως μικρότερες ανάγκες, αλλά σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια, ε, τα αιτήματα θα έλεγα, οι προσδοκίες παραμένουν στο ίδιο ε, επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πρασπιστούμε τις δυνατότητες που έχουμε. Επίσης αναφερθήκατε στα καταπιστεύματα. Τα καταπιστεύματα είναι αρκετά ικανά μέσα για συγκεκριμένες δράσεις. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με ε, τακτική, αν αναφορά και παρουσίαση της χρήσης των κονδυλίων από τα καταπιστεύματα. Η πρώτη έκθεση, αν δεν έχει ακόμα αποσταλεί, θα αποσταλεί άμεσα και νομίζω ότι υπάρχει, είναι σαφές, ε, το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετέχει και στα διοικητικά συμβούλια των καταπιστευμάτων και να αντιπροσωπεύεται σε αυτά. Ένα τελευταίο σημείο για μας. Ε, χαιρετίζουμε χθε ότι υπήρξε μια ψηφοφορία ανάμεσα στις επιτροπές, της αρμόδιες, και θα προχωρήσουμε ιδιαίτερα στο ερώτημα το οποίο τέθηκε προβλέπεται για τον προϋπολογισμό του 2018 το λεγόμενο replenishment, η ανατροφοδότηση. Και προβλέπεται επίσης ότι οι συνεισφορές του ΦΕΔ να δοθούν κανονικά το 2018. Δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω στην παρούσα φάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Μουρεσάν, θέλετε να αντιδράσετε και μετά θα δώσω το λόγο στον ε, Γκέρενς. Δεν θα σας καθυστερήσω άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Γκέρενς, ε, συμφωνώ μαζί σας, η συνοχή είναι σημαντικό αυτό, το βλέπουμε αυτό τον επισκεπτόμεθα τις χώρες. Δεν μπορούμε εμείς να αναφερθούμε στις βασικές αιτίες ε, της μετανάστευσης, αν δεν βρούμε λύσεις σε με τις ανάγκες των πληθυσμών στον τομέα των υποδομών, της κατοικίας, της εκπαίδευσης, της υγείας, αν δεν υπάρχει σταθερότητα από πλευράς μας. Για τα trust funds, τα καταπιστεύματα, να πω ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θεωρεί τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν ε, τα καταπιστεύματα ως εξής, δηλαδή κάτω από πιεστικές καταστάσεις, κατεπίγουσες ανάγκες, δεν υπήρχε ίσως άλλος τρόπος να προσθέσουμε ε, κάτι ε, στην κάλυψη των αναγκών αυτών. Η συμμετοχή του Κοινοβουλίου είναι πραγματικά απαράδεκτη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου θα πρέπει να διασφαλιστούν, θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ενότητα του προϋπολογισμού και ουδέποτε εμείς ε, θα συνηθίσουμε στην ιδέα να μαθαίνουμε από τον τύπο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίδει χρήματα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό ενώ η ε, ε, συναρμόδια αρχή επί του προϋπολογισμού δεν έχει ιδέα. Συνεπώς λοιπόν τα πράγματα θα πρέπει να μπουν σε μια κάποια τάξη και να σταματήσουμε πλέον το κοινοβούλιο ε, να αγνοείται. Τώρα για το Brexit, σημαντικά αυτά τα οποία είπατε κύριε Γκέρεντς όπως και οι άλλοι συνάδελφοι. Εγώ είμαι υπεύθυνο για το 2018 και θα πρέπει να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει Brexit για το 2018. Δεν υπάρχουν συνέπειες λοιπόν. Το 2018 το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι μέλος της Ένωσης με πλήρη δικαιώματα και πλήρης ευθύνες. Συνεπώς λοιπόν δεν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικές προκλήσεις. Όμως θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο εργαζόμεθα και δυστυχώς χάνουμε ε, ένα κράτος μέλος, ε, χάνουμε έναν καθαρό συνεισφορέα ο οποίος προσέφερε στον προϋπολογισμό και απαιτείται να βρεθεί μια μακροπρόθεσμη λύση. Εμείς στην Επιτροπή Προϋπολογισμών δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στους ιδίους πόρους και ο τρόπος με τον οποίο θα καθοριστούν στο μέλλον έτσι ώστε να μην επιβαρύνουν τον Ευρωπαίο πολίτη αλλά από την άλλη να μπορέσουν και να ανταποκριθούν σε μια πιο προβλέψιμη δημοσιονομική κοινοτική πολιτική και να αποφύγουμε τα παζάρια ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα στα πλαίσια της απόφασης για το νέο δημοσιονομικό Τώρα επίσης και η αλλαγή επίπεδου και για την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, Τράπεζα Επενδύσεων μάλλον, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ είμαι σκιώδης για τα θέματα αυτά της ομάδας μου. Απαιτούνται 30 δις εδώ για να υπάρξει αναβάθμιση αυτή. Νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο επίπεδο προσδοκιών. Νομίζω όμως ότι οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο εδώ θα είναι πολύ σκληρές για να κλείσουμε. Λοιπόν, έχουμε νέες προτεραιότητες, δεν τις είχαμε προβλέψει στην αρχή του πολιετούς δημοσιονομικού το 2013. Οι νέες αυτές όμως προτεραιότητες δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τα υπάρχοντα, τα προσχεδιασμένα και τα μελλοντικά μας προγράμματα. Ε, κατανοώ αυτό που είπε και η κυρία Χάουταλα, ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην άμεση γειτονία, διότι από εκεί προέρχονται οι περισσότερες προκλήσεις. Κοιτάξτε, το θέμα της εκρίζωσης της φτώχειας είναι γενικό. Σαφώς δεν θα πρέπει να αγνοούμε τις νέες προτεραιότητες, αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοούμε τα ισχύοντα και τρέχοντα προγράμματα. Για να καλύψουμε τις νέες ανάγκες απαιτούνται νέοι πόροι και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διευκρινίσει στην ολότητά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν η Ένωση καλείται να κάνει περισσότερα, είναι σαφές ότι θα υπάρξουν ανάγκες και για νέους πόρους, όπως είπαν και κάποιοι από εσά. Λοιπόν, αυτά συνάδελφοι, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ε, εγώ είμαι απολύτως διαθέσιμος για να ακούσω τις απόψεις σας για την τρέχουσα διαδικασία του προϋπολογισμού και όπως είπα μην ξεχνάτε την 3η Μαΐου σαν πλαίσιο προθεσμία για να στείλετε τις απόψεις σας. Σας ευχαριστώ για την ευκρίνεια της παρουσίασής σας. Συμφωνούμε με αυτά τα οποία είπατε νομίζω. Ο κύριος Γκέρντς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινώ με μια διαπίστωση. Όλοι συμφωνούμε, το είπα στην αιτιολογική έκθεση, ότι είμαστε ομόφωνοι ως προς τις μεγάλες προτεραιότητες και αυτό που θα πρότεινα υπό τη μορφή ψηφίσματος στο κοινοβούλιο μου μας. Ο Βασάν αναφέρθηκε σε πολλά σημεία και θα επανέλθω σε αυτόν να πω ότι το 20% τον ε, του προπολογισμού θα πρέπει να πάει στι ε, αναπτυσσόμενε, λιγότερο αναπτυγμένε χώρε. Συμφωνώ, Βινσάν, με όλα όσα είπε. Η Χάιντι Χάουταλα θύμισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε με την ε, διοργάνωση της ασφάλειας και το χρηματοδότηση αντίστοιχα από το προϋπολογισμό. Να θυμίσω ότι η ασφάλεια είναι μία έννοια πιο ευρεία από την αστυνομική ή στρατιωτική παρέμβαση. Υπάρχει ασφάλεια της απασχόλησης, διατροφική ασφάλεια, κοινωνική ασφάλεια. Αυτοί οι τομείς είναι στη δική μας αρμοδιότητα και είναι αυτές ε, που λιγότερο τελικά εποπτεύονται. Ε, και υπάρχει ε, μεγάλη χρηματοδότηση προς την καταστολή, προς ε, τον ε, στρατό, την αστυνομία και την εξωτερική ασφάλεια. Όταν οι σειράξεις είναι εμφύλες περισσότερο και όχι τόσο... Και δεν είναι πλέον τόσο εμφύλες αλλά είναι διεθνείς και υπάρχει και υποβόσκουσα η φτώχεια, θα πρέπει εμείς να ενσκύψουμε και να μην ε, ξεχνάμε ότι ε, αυτή η μάχη είναι μια μάχη όχι μόνο για την ασφάλεια αλλά και την εκρίζωση της ε, φτώχειας. Επίσης, να σας θυμίσω, το Παγκόσμιο Ταμείο για το AIDS, την φυματίωση και τη μαλάρια χρηματοδοτείται για να μπορέσει να επιλύσει μεσοπρόθεσμα προβλήματα με διάφορες μορφές ε, πόρων από τα κρατημέλη, από την Κομισιόν, από τον Bill Gates, από μη κυβερνητικέ οργανώσεις, από ιδιωτικά ιδρύματα. Ε, αν δεν υπάρχει προβλεψιμότητα και αν σταματήσουμε ή μειώσουμε τη χρηματοδότηση, καταδικάζουμε σε θάνατο αυτούς που επωφελούνται από μία ε, θεραπεία για το AIDS, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να διατηρήσουμε την προβλεψιμότητα. Συμφωνώ κύριε Βαντά για την ε, πολύ αποφασιστική ε, υπεράσπιση του 0,7%. Ελπίζω να το κάνουμε σε όλους τους τομείς και μέσα στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου που έχουμε αυτή τη στιγμή με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Ξέρω ότι αυτό το πράγμα θα, μας, ε, θα είναι σπαζοκεφαλιά για μας μέχρι τα τέλη των διαπραγματεύσεων. Η Αν Λίτς ε, πήγε προς την ίδια ο Αν Λίτς πήγε προς την ίδια κατεύθυνση. Ε, ξέρουμε σε τι βαθμό έχει φτάσει για να πείσει τη χώρα του να περάσει αυτό στο εκλογικό πρόγραμμα. Έκανε τα πάντα. Και μια τελευταία λέξη τώρα για την έξοδο της ε, Βρετανίας. Είπαμε ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε μεταξύ μας ε, για το πώς θα κάνουμε τις προτάσεις. Ε, πρέπει να το συζητήσουμε γιατί έχουμε όλες οι ιδέες, ιδέες και πρέπει να έχουμε μια δομημένη προσέγγιση, να δούμε πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε. Ένα όμως είναι σίγουρο. Όταν φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα χρηματοδότησης, όχι μόνο στα πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής λόγω της έλλειψης της τεχνογνωσίας από την Βρετανία, αλλά θα υπάρχει και μια μάχη μεταξύ όλων των τμήματων σχετικά με τα κονδύλια ε, που θα πρέπει ε, να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις θέσεις του 1%. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ε, ότι θα υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ της ΚΑΠ, των διευθυντικών ταμείων, της ανθρωπιστικής βοήθειας ε, για το πώς θα διαρθρωθούν τα κονδύλια. Η Κομισιόν είναι σε άλλη γραμμή σε τέτοιο βαθμό που είμαι σίγουρος ότι με την Κομισιόν μπορούμε να κάνουμε ένα μπλοκ ενάντια στους τσιγκούνιδες του Συμβουλίου. Για να δούμε τι θα γίνει στις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι καλύψαμε τα βασικά σημεία. Σάρλ, ε, τώρα για τα πιλωτικά προγράμματα Προθεσμία είναι την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω ότι θα στείλετε κάτι στους συντανιστές σήμερα ή αύριο ε, και θα τους ε, ζητήσετε να στείλουν τα project μέσα στην προθεσμία. Επίσης ζητήσαμε από τους συναδέλφους να στείλουν project τα οποία θα πάνε στην Κομισιόν για να ελεγχθούν, ε, τα οποία θα είναι καλά. Ήδη το έχουμε κάνει αυτό, έχει γίνει. Οπότε, θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι είναι καλά τα project αυτά και ότι δεν θα σπαταλήσουμε τον χρόνο της Κομισιόν. Λιγότερα και πιο ποιοτικά πιλωτικά προγράμματα χρειαζόμαστε για την επιτροπή μας. Μετά την παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισμού τέλη Μαΐου, η δική μας επιτροπή θα απαντήσει, ο κύριος Γκέρενς ε, θα συντάξει επιστολή και μετά αργότερα γνωμοδότηση που θα ψηφιστεί στην πρώτη συνάντηση μετά τις ε, θέρινες διακόπες. Σας ευχαριστώ όλους. Νομίζω ότι η συζήτηση ήταν πολύ χρήσιμη και επικοδομητική. Ευχαριστούμε κύριε Μωρισόν. Δεν ξέρω αν θα σας ξαναδούμε ε, σύντομα μετά από αυτή την μακροσκελή διαδικασία για τον προπολογισμό. Πάμε στο σημείο 14. Δημιουργία εργαλείου που θα συμβάλλει στη σταθερότητα και στην ειρήνη. Εύκολο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι απάντηση της Επιτροπής μας στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός εργαλείου που θα συμβάλλει στη σταθερότητα και την ειρήνη. ICSP. Ε, αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και συνεργαζόμαστε με την ΑΦΕ, την Επιτροπή, βάσει του κανόνα 53 συν ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών. Η Επιτροπή μας ήθελε να έχει μεγαλύτερο λόγο για την εξέλιξη αυτού του φακέλου, αλλά δεν κέρδισαμε αυτή τη μάχη. Δεν πειράζει, έχουμε ένα εξαιρετικό εισηγητή που θα μας παρουσιάσει τη γνωμοδότησή του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Λίντα. Δεν ξέρω αν θα είναι εύκολο το εγχείρημά μου. Πολύ αμφιβάλλω. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μια πρόταση. Και η ιδέα είναι να συμπεριληφθεί ένα νέο άρθρο που θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διευρύνει τα συστήματά της υπό επίγουσες συνθήκες στη δυνατότητα στην, ώστε να μπορεί να βοηθά τους εταίρους να αποκτούν δυνατότητες σε στρατιωτικό και άλλο σκέλος προς όφελος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στις χώρες τις οποίες βοηθά αναπτυξιακά. Αρμόδια Επιτροπή είναι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και ο κ. Ντανσάν είναι εκεί ο εισηγητής. Στο σχέδιο γνωμοδότησής μου έχω περιορίσει τις προτάσεις μου σε πέντε τριοτροπολογίες, πολύ συγκεκριμένες, πολύ απλές και ευθείες, ειλικρινείς βασική τροπολογία στο σχέδιο γνωμοδότησης είναι η τροπολογία 4. Θέλουμε να υπάρχει μια νέα διάταξη που ε, θα μπει στο ICSP και θα λέει ότι οποιαδήποτε δράση για την απόκτηση ε, τέτοιων δυνατοτήτων από αυτούς τους λαούς θα εκπληρούνται με τα κριτήρια του ε, Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη και έχουμε και τις ανα, αναθεωρημένες ε, οδηγίες ε, του ΟΣΑ. Χρησιμοποιούμε ακριβώς ε, τη διατύπωση του σχετικού κανονισμού. Η πρόταση εκφράζει τις ανησυχίες μας για τα θέματα διαφάνειας, λογοδοσίας, για το capacity building, για τη ε, στήριξη και την ανάπτυξη σε ευάλωτες χώρες και σε χώρες που ε, ε, είναι αποσταθεροποιημένες και αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Στόχος είναι η μείωση και σε βάθος χρόνου εξάλληψη της φτώχειας. Εξέφρασα αμφιβολίες για το είδος της αποστολής μας, γιατί είχα υπόψη μου το σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Ντανσάν. Ε, χθες το έλαβα. Βλέπω ότι έχει συντάξει την πρόταση που υποβάλλει στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και εντωμεταξύ έχει συμπεριλάβει ριζοσπαστικές αλλαγές στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλώς προτείνει περιορισμένη χρηματοδότηση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων σε κατεξαίρεση συνθήκες και περιστάσεις. Ο κ. Ντανσάν τώρα προτείνει πολύ ριζοσπαστικές αλλαγές σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην τροπολογία υπαριθμών 3, το όρος exceptional θα πρέπει, ε, θα πρέπει να αντικατασταθεί με τον όρο specific, ειδικέ, συγκεκριμένες, ιδιαίτερες. Το exceptional βεβαίως είναι πιο ισχυρό ως όρος. Ε, αλλά, το, αλλά επιδέχεται περισσότερων ερμηνεών. Έχουμε την τροπολογία 5, όπου ο κύριος Ντανσάν θέλει να διαγραφεί η λέξη ανάπτυξη, να αφαιρεθεί. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η βοήθεια μπορεί να καλύψει ιδιαίτερο στην διάταξη των προγραμμάτων χτισήματος δυνατοτήτων σε, για θέματα σταθερότητας και ανάπτυξης. Και θέλει ο κ. Ντανζάν να διαγραφεί αυτή η τελευταία λέξη και ανάπτυξης. Και έχουμε τις τροπολογίες 7 και 8 που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή τονίζει ότι οι κατεξαίρεσεις περιστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, στην πρώτη παράγραφο, θα πρέπει να ε, αναγυγνώσκονται με σωρευτικό τρόπο. Παράγραφος 3, ε, εδάφιο Α και Β, θα πρέπει αυτά να διαβάζονται από κοινού, να ερμηνεύονται από κοινού και να εκπληρώνονται όλα αυτά από κοινού για να ισχύουν. Τώρα ο κύριος Τανσάν προτείνει στο τέλος του σημείου α να αντικατασταθεί η λέξη και με τη λέξη ίδια ζευτικό. Και τέλος, επιπρόσθετα στο σημείο β, θα ήθελε ο αρμόδιος από την Επιτροπή ΑΦΕΤ να αλλάξει τη διατύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία λέει ότι όπου υπάρχει συνένεση μεταξύ της ενδιαφερόμενης χώρας και της διεθνούς κοινότητας και ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεξής, τέλος της παράθεσης, θέλει ο κύριος Ντανσάν να ε, διαγραφούν οι λέξεις διεθνούς κοινότητας. Άρα, να, αν διαβάσει κανείς την πρόταση του κυρίου Ντανσάν, στο σύνολό της βλέπει ότι μπορεί κανείς να αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο χρηματοδότηση σε περιστάσεις όπου υπάρχει συνένεση μόνο μεταξύ της ενδιαφερόμενης χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς άλλες προϋποθέσεις ή ε, προπετούμενα. Αυτή είναι μια πολύ ριζοσπαστική αλλαγή που προτείνει ο κ. Ντανσάν. Λοιπόν, Εμείς έχουμε τη γνωμοδότησή μας για το σκέλος της αναπτυξιακής πολιτικής που έχει να κάνει με τον κανονισμό και περιμένω τροπολογίες από τις πολιτικές ομάδες και με χαρά θα συζητήσω με τους σκιώδες εισηγητές για τη γνωμοδότησή μας. Και πρέπει να δούμε πώς θα προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την Επιτροπή ΑΦΕΤ, όταν εγκρίνει το τελικό ε, σχέδιο έκθεσης. Αυτά λοιπόν θα ήθελα να πω αρχικά ως εισαγωγικέ παρατηρήσεις και με χαρά θα ακούσω τα σχόλιά σας και ε, περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να έχουμε στενή συνεργασία. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Σας ευχαριστούμε πολύ μετά από αυτά που ακούσαμε να μας λέτε για την ΑΦΕΤ. Ο κύριος Βέντε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, ομιλώ εκ μέρους του κύριου Πόγκα για άλλη μια φορά γιατί είναι ο σκιώδη για το ΕΛΚ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του ο άξονας ασφάλειας και ανάπτυξης είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών μας τα τελευταία χρόνια. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος η ασφάλεια είναι συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και καλωσορίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ ασφάλειας και ανάπτυξης και για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ε, των πολιτικών ασφάλειας και πολιτικών ανάπτυξης, κυρίως στις χώρες όπου υπάρχουν ε, συγκρούσεις και περιοχές που υπάρχουν συγκρούσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει το παν για να διασφαλίσει την αξιοπιστία της εξωτερικής μας δράσης και κυρίως την εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών σε βάθος χρόνου, με προοπτικές μακροχρόνιες. Θα συμβάλλουμε στο σχέδιο οκνομοδότηση, θα υποβάλουμε τροπολογίε και θα συνεργαστούμε στενά με τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γερμανικά πολύ για την εργασία ε, που έκανε ο εισηγητής. Ε, έχω εμπλακεί σε αυτό το θέμα με πολλούς τρόπους, γιατί η Επιτροπή, ε, γιατί είμαι μέλος όχι μόνο της Επιτροπής για την Ανάπτυξη, αλλά και της ΑΦΕΤ. Θεωρώ ότι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής που έχει να κάνει και με την πολιτική ασφάλειας, είναι πολύ σημαντικό να εισάγουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Θεωρώ ότι πρέπει εκ των προτέρων να δούμε πώς ε, θα το δομήσουμε αυτό ε, δημοσιονομικά. Πρέπει εκ των προτέρων να δούμε ε, ποια είναι η σημασία της πολιτικής ανάπτυξης και του ε, προϋπολογισμού για την ε, στόχους ε, της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει εκ των προτέρων να δώσουμε ένα τίμημα λοιπόν για αυτούς τους στόχους. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι και στη Γερμανία έχει γίνει το ίδιο. Υπάρχει μια γραμμή του προϋπολογισμού στο Υπουργείο Άμυνας. Είναι το σχέδιο του προϋπολογισμού που δίνει 130 ε, εκατομμύρια ε, ευρώ ως security instrument. Είναι λίγο διαφορετική διατύπωση, όμως ακριβώς αυτό κάνει. Είναι εργαλεία για την ασφάλεια, για την ε, ενίσχυση των missing links, των στοιχείων που λείπουν ώστε να ενισχύσουμε την ασφάλεια και εμείς εδώ ως ε, Κοινοβούλιο λαμβάνουμε εδώ έναν νέο προϋπολογισμό στον οποίο υπάρχει μια επίθεση προς τον προϋπολογισμό της ανάπτυξης και πρέπει να είμαστε πολύ συνεκτικοί ως προς την προσέγγιση μας ε, για να μην έχουμε ε, προβλήματα τελικά να δούμε πώς θα μπορέσουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις να συνεργαστούν με τους ε, οργανισμούς άμυνας, να υπάρχει μια ενίσχυση αυτή της συνεργασίας, ε, όμως αυτό να ενισχυθεί ε, όχι μόνο ως ε, μια γραμμή της αναπτυξιακής πολιτικής, αλλά ως μια χωριστή γραμμή. Η Επιτροπή έχει συνεργαστεί με τον ΩΣΑ και έχει διευρύνει τα στάνταρ ασφάλειας και ε, όλα αυτά τα θέματα σχετίζονται μεταξύ τους, οπότε θα πρέπει να τα εξετάσουμε πιο στενά. Ευχαριστώ. Είναι κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει να λάβει το, λόγο. Αν όχι, έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις για την Κομισιόν. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο πολύ για πόσα χρήματα μιλάμε σε αυτό το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο και από πού έρχονται τα χρήματα στο προϋπολογισμό. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Συνεχώς μου λένε ότι υπάρχει προβλήματα προβλήματα ε, στην Κομισιόν. Έχουν ζητηθεί κάποιες αλλαγές. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα με τα αναπτυξιακά κονδύλια ε, σε αυτό το νέο εργαλείο. Μπορείτε να μας το διευκολύνετε γιατί έχουμε φτάσει σε έναν διάλογο και θεωρούσαμε ότι το πρόβλημα είναι μόνο το exceptional αλλά τελικά είναι άλλα πέντε πράγματα. Ε, ποια είναι η άποψη. Ξέρω ότι το Συμβούλιο έχει μια κοινή θέση και είναι το ε, δεν είναι εδώ το Συμβούλιο και η Κομισιόν δεν ξέρει ποια είναι η θέση του Συμβουλίου. Οπότε ίσως να σας δώσω το λόγο. Έχουμε τον Ρούντι Σάλτς εδώ, το Γενικό Διευθυντή. Να του δώσω το λόγο να μας απαντήσει ίσως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια επικοδομητική και χρήσιμη ε, γνωμοδότηση. Δεν μπορώ να κάνω σχόλια για τις ε, προτάσεις της ΑΦΕΤ. Κάποιες έχουν να κάνουν με το Συμβούλιο. Εμείς υποστηρίζουμε τη θέση του Συμβουλίου και θέλουμε ακόμα να περιμένουμε λίγο μέχρι να κάνουμε τα σχόλια για τη θέση της ΑΦΕΤ. Να πω όμως κάποια πράγματα σκεφτικά Νομίζω ότι ε, αυτό το θέμα έχει να κάνει με την πρόταση ε, που έκανε το Συμβούλιο στην Κομισιόν να βρει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα είναι ευρύτερο από αυτό που έχουμε εδώ. Αυτό που πρότεινε τελικά η Κομισιόν είναι μια ελάχιστη τροποποίηση του ICSP, το διεύρυνε ακριβώς στα σημεία που ο κύριος Βάριεν ανέφερε προηγουμένως, γιατί υπάρχει ένα σημείο που λείπει εδώ από την εργαλειοθήκη μας. Ε, ε, την εργαλειοθήκη των εργαλείων για την ασφάλεια και την ανάπτυξη και βρισκόμαστε στο όριο μεταξύ ε, ασφάλειας και ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν η τροποποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών του ΩΣΑ ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη όμως οι κατευθυντηρίες γραμμές του ΩΣΑ δεν έχουν σχεδιαστεί για να θεσπίζουν πολιτικές. Εμείς, εσείς και το Συμβούλιο το κάνουμε αυτό. Τα πράγματα λοιπόν που προτείνουμε για να μπορέσουμε να τα επιτύχουμε μέσω του ICSP ε, είναι δεν, δεν έχει σχεδιαστεί έτσι αυτό το εργαλείο. Πραγματικότητα είναι ότι τα περισσότερα από αυτά που κάνουμε στο ICSP έχουν αυτή την ιδιότητα και ίσως οι συνάδελφοι θα μπορούσαν να ε, μας ε, το αναφέρουν αυτό. Και όταν μιλάμε για την ε, ασφάλεια και τη σταθερότητα με μέσα πολιτικά, μπορούμε να το κάνουμε. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα χρήσιμο, μια χρήσιμη εργαλειοθήκη και υποστηρίζουμε την γνωμοδότηση, το μόνο σημείο που πραγματικά δεν μπορούμε, με το οποίο δεν μπορούμε να συμβαδίσουμε είναι αυτό το θέμα του κατά πόσο είναι το ICSP. Δεν είχε σχεδιαστεί έτσι. Ε, το άρθρο 3α μπορεί να είναι, αλλά πρέπει να το ξέρουμε αυτό εκ των προτέρων. Επειδή δεν το ξέρουμε, ε, θα το ξέρουμε όταν θα διαμορφωθούν οι επιχειρήσεις Θα δούμε αν θα είναι το ή όχι. Είμαστε στα όρια ε, της ασφάλειας αλλά όχι της ανάπτυξης. Με τη νέα αναπτυξιακή ατζέντα η ανάπτυξη έχει έναν ορισμό, ο οποίος τώρα ε, περιλαμβάνει την προώθηση της ειρηνικής βιώσιμης κοινωνίας ε, ε, στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του 2014. Τα συζητήσαμε αυτά στη συνένεση. Σκεφτόμαστε μέσα στα πλαίσια ενός νέου πλαισίου πολιτικής και ακριβώς γι' αυτό τον λόγο θεωρούμε ότι Μπορούμε εδώ να κάνουμε κάποια πράγματα με αυτό το εργαλείο τα οποία συνεισφέρουν στην ανάπτυξη. Ο πρωταρχικός στόχος πρέπει πάντοτε να είναι η ανάπτυξη και γι' αυτό θεωρούμε ότι έχουμε σεβαστεί και την πολιτική καθοδήγηση σε αυτό τον τομέα. Τώρα για τα πιο συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν. Τα χρήματα για αυτήν την τροποποίηση, όπως ξέρετε, προβλέψαμε όχι πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για την εναπομείνασα περίοδο του προϋπολογισμού. Στην ουσία, αυτά θα πάνε από τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΑ, από το αποθεματικό, από το εργαλείο για τη γειτονία και από το εργαλείο για την ανάπτυξη, περίπου σε ίσα μέρη. Ε, όσο περισσότερα χρήματα ε, δίνουμε, τόσο περισσότερο ε, ντάκαμπλ θα γίνονται. Τώρα, να απαντήσω στα δικά σας ερωτήματα, Πρόεδρε. Νομίζω ότι ε, ήμασταν ξεκάθαροι σε αυτό και αν μου επιτρέπετε να δώσω τα... στο συνάδελφο το λόγο για να σας πει τι κάνουμε στο ICSP και πώς θα ε, αντιμετωπίζουμε το θέμα του Dacability. Ευχαριστώ. Όπως είπαν ε, ήδη οι συναδελφοί, το εργαλείο αυτό δεν ε, δεσμεύεται άμεσα από κριτήρια αναπτυξιακής ενίσχυσης. 90% των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από το εργαλείο αυτό είναι Dacable. είναι ε, τώρα κάτι που δεν έχει να κάνει με την επίσημη ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Υποστηρίζουμε διάφορες ε, πτυχές μιας αποστολής παρακολούθησης. Αυτό που κάνουν οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί είναι προϋπόθεση για την σταθερότητα στην περιοχή, αλλά δεν είναι επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια αυστηρά. Το κέντρο της βαρύτητας της πρότασης της Κομισιόν είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας εταίρου. Όπως είπε ο συνάδελφος λοιπόν, αυτή η πρόταση είναι, ξεκάθαρα, είναι ξεκάθαρη. Έχει κάποια ξεκάθαρα όρια. Θέλει να φέρει ένα επιπλέον στοιχείο στην εργαλειοθήκη το οποίο ε, υπάρχει για πολύ συγκεκριμένες εξαιρετικές περιστάσεις. Ευχαριστώ. Να κάνω μια ερώτηση. Να μας δώσετε ε, ένα παράδειγμα. Ε, είπατε κάτι για την Ουκρανία, αλλά είναι λίγο... Είναι υπό εργαλείο αυτό. Εδώ προτείνετε ένα νέο εργαλείο. Θέλετε ένα νέο εργαλείο για να κάνετε κάτι διαφορετικό. Αν παίρνετε 25% DCI ε, της αναπτυξιακής ε, βοήθειας δηλαδή του DCI, παίρνετε αυτά τα χρήματα από το ένα μέρος και τα πάντε σε ένα άλλο. Αυτοί οι κανόνες που εφαρμόζονται για το DCI εφαρμόζονται και σε αυτό, όχι. Καταλαβαίνω λοιπόν το θέμα σας, αλλά μάλλον πρέπει να βρούμε μια λύση γι' αυτό. Τα κράτη-μέλη που αναφέρουν την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, το λένε στην Κομισιόν. Η Κομισιόν λέει στα κοινοβούλια τους, ε, αυτό είναι επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Αν τα βγάλετε από τον κορβανά αυτόν, πώς θα την αναφέρουν. Αυτό είναι το θέμα. Κύριος Γκέρενς. Να επανέλθω σε αυτό το θέμα που θέσατε. Δεν ξέρω αν το παράδειγμα που δώσατε είναι το καλύτερο σύμφωνα με την αρχή της διαφοροποίησης η Ουκρανία δεν θα πρέπει να παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε από αυτή την άποψη η υπόθεση αυτή δεν ισχύει. Είχαμε μία συζήτηση προηγουμένως για το θέμα της ασφάλειας. Υπάρχει ένα κομμάτι προληπτικό, ένα κομμάτι αναπτυξιακό και ένα κομμάτι κατασταλτικό. Υπάρχουν μάλιστα και ορισμένες χώρες οι οποίες στα πλαίσια των ανακοινώσεών τους για την βοήθεια προς την ανάπτυξη αρνούνται να συμπεριλάβουν ε, ορισμένες δράσεις οι οποίες είναι duckable και οι οποίες είναι συμβατές ε, με την Επιτροπή του ΩΣΑ. Ε, πολλές είναι οι χώρες αυτές, Σουηδία και η δική μου χώρα, αρνείται να συμπεριλάβει στις ετήσιες δημοσιεύσεις στοιχείων τις συνεισφορές που δόθηκαν προς τους πρόσφυγες την πρώτη χρονιά υποδοχής. Δεν είμαστε ε, υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε λοιπόν το περιθώριο το οποίο προβλέπει για τις χώρες η Επιτροπή για την Ανάπτυξη του ΩΣΑ αν θέλουμε να αποδείξουμε το αντίθετο μέσω του παραλόγου, αν θέλουμε πραγματικά να καταργήσουμε το χρέος ας πούμε, μπορούμε να διαθέσουμε το σύνολο του προϋπολογισμού στην κατάργηση του χρέους, οπότε σε αυτή την άποψη δεν θα είχαμε κάνει τίποτα σε επίπεδο αναπτυξιακό, αλλά φυσικά θα είχαμε καλύψει 100% τις ανάγκες της Επιτροπής για τη βοήθεια για την ανάπτυξη. Αν δανείσετε ένα δις στον Μομπούτου σαν παράδειγμα, δεν σας έχει επιστρέψει ούτε ένα ευρώ, γέμισε τις τσέπες του και ο, ο Μπερνάρ Κουσνέρ είχε πει ότι ο Μομπούτου ήταν ένας, ένα χρηματοκιβώτιο αυτοκινούμενο και φόραγε και ένα καλπάκι από δέρμα λεοπάρδαλης. Λοιπόν, ε, ε, πέραν αυτού τίποτα. Λοιπόν, πρέπει εμείς να χρησιμοποιούμε το σύνολο των περιθωρίων που μας δίνει η Επιτροπή του ΩΣΑ. Θα δώσω το λόγο πάλι στον κύριο Βάιρεν. Η Αν έχει ζητήσει όμως ξανά το λόγο. Κοιτάξτε, έχουμε το ίδιο ακριβώς ε, μέσο και στην Γερμανία. Γιατί λοιπόν δεν είναι δυνατό να έχουμε μια νέα γραμμή και να έχουμε συγκεκριμένα μέσα τα οποία να είναι εντάκαμπολ. Υπάρχει ένας κατάλογος ε, των καταστάσεων οι οποίες καλούνται να καλυφθούν από τις κυβερνήσεις όπως ο έλεγχος ε, των συνόρων σαν παράδειγμα. Το θέμα της ασφάλειας στις διάφορες χώρες που παίρνουν βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό ίσως θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα γραμμή η οποία οποία θα αντικατοπτρίζει την πραγματική συνοχή. Το να λέμε ότι έχουμε μια συνοχή, συνεκτική πολιτική δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης στη Γερμανία δεν θα ήθελε να υπάρξει η δυνατότητα για να χρησιμοποιείται η αναπτυξιακή βοήθεια για θέματα ασφάλειας, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών σκοτίστηκε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει λίγο να το διευκρινίσουμε αυτό καλύτερα για να δούμε αν μία κάποια παρέμβαση είναι ντόκαμπολ ή όχι. Εγώ δεν είμαι απόλυτα πεπισμένος στην παρούσα φάση. Φαίνεται ότι έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες. Ας πούμε, αν από τα 100 εκατομμύρια πάρουμε τα 25 από το DCI, δημιουργούμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Ίσως την επόμενη φορά να μπορέσει κανείς περισσότερα χρήματα να πάρει από το DJI. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ε, τι γίνεται ε, ε, με το ODA. Χάνουμε και το 0,7. αν θέλετε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο μέσο δεν έχετε παρά να το δημιουργήσετε και να καλύψετε τις δημοσιονομικές ανάγκες αλλά δεν χρειάζεται να φωνάζουμε ότι θέλουμε κάτι και να μην κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι όταν παίρνουμε χρήματα από τη μία γραμμή αυτό δεν θα πρέπει να λειτουργεί εις βάρος της γραμμής αυτής και γι' αυτό όταν ε, καθορίζονται κάποιες χρήσεις πιστώσεων θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η χρήση αυτή. Οι ερωτήσεις σας είναι πολύ δικαιολογημένε. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς είναι θα έλεγα μια βραχυπρόθεσμη απάντηση σε ένα ευρύτερο αίτημα του Συμβουλίου. Επιλέψαμε να το κάνουμε αυτό γιατί για το παρόν δημοσιονομικό πλαίσιο Έχουμε τα μέσα στον τίτλο 4, μεταξύ των οποίων το ISP. Και αυτό το οποίο προτείνουμε εδώ είναι κάτι το οποίο θεωρείται ότι θα ήταν καλύτερα να διευρύνουμε λίγο το, ISP, το οποίο έχει μια συγκεκριμένη θέση στον προϋπολογισμό το ICSP λοιπόν έχει μια ξεκάθαρη εντολή, πολύ ευρύτερη από αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, οπότε θα μπορούσαμε να κατανείμουμε τη γραμμή του προϋπολογισμού που έχει στη διάθεσή του με το σωστό τρόπο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ουσιαστικά. Χρησιμοποιούμε ένα υπάρχον μέσον το οποίο είναι πρόσφορο και εκεί βάζουμε χρήματα από διαφορετικές πηγές και το κάνουμε αυτό γιατί αναγνωρίζουμε ακριβώς ότι δεν είναι μόνο ανάπτυξη, δεν είναι μόνο ασφάλεια και θα δούμε στα πλαίσια του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου, ε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ε, μια πρόταση για ένα νέο μέσο ασφάλειας στο εσωτερικό του προϋπολογισμού της. Αυτό είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να γίνει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θέλει, λέει, να αυξήσει το ρόλο της σε επίπεδο προβλημάτων διεθνών στον τομέα της ασφάλειας. Λοιπόν, το θέμα εδώ είναι σχετικά περιορισμένο. Κληθήκαμε εμείς να ανταποκριθούμε και χρησιμοποιούμε ένα υπάρχον μέσο, γιατί ήδη το κάνει αυτό το συγκεκριμένο μέσο. Απλά δεν μπορεί να κάνει κάποια άλλα πράγματα τα οποία ζητούν κάποια χρήματα να πηγαίνουν στους βασικούς χρήστες απευθείας. Το να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα εντελώς νέο μέσο και μια εντελώς νέα γραμμή ε, του προϋπολογισμού για να ανταποκριθούμε στο αίτημα του Συμβουλίου δεν θα είχε νόημα. Εν πάση περιπτώσει αυτή είναι μια συζήτηση η οποία θα πρέπει να ξαναγίνει. Να απαντήσω και σε κάτι που είπε ο κύριος Βάιριναν προηγουμένως και ίσως ξέχασα να απαντήσω. Το ICSP είναι διαφανέστατο. Υπάρχει επίσης κάθε ε, τρεις μήνες μια έκθεση των δράσεων που χρηματοδοτούμε και μπορεί κανείς να είναι βέβαιος για το τι κάνουμε ακριβώς και πώς το κάνουμε. Συνεπώς η διαφάνεια αυτή εγγράφεται από την ε, ε, τριμηνιαία έκθεση για τα οικονομικά του ICSP. Ο εισηγητής του σχεδίου γνωμοδότησης. Ευχαριστώ. Η καλύτερη λύση είναι η λύση του κυρίου Αναλίντς. Να υπάρχει μια γραμμή στο προϋπολογισμό στο πλαίσιο του CSFP που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς και να δημιουργηθεί. Μέρος αυτής της χρηματοδότησης θα μπορούσε να είναι επιλέξιμο βάση του DAC, δηλαδή να αναφέρεται στον ΩΣΑ και δεν θα είχα μεταφορά χρημάτων από το DCI σε αυτή τη γραμμή του προϋπολογισμού. Νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή λύση. Άλλη λύση είναι να έχουμε μια γραμμή του προϋπολογισμού στο CSFP και πέρα από αυτή τη χρηματοδότηση να αξιοποιήσουμε ε, χρηματοδότηση αναπτυξιακή, DCI. Για πρακτικούς λόγους όμως το λογικό για μένα είναι να έχουμε ένα εργαλείο που θα έχει χρήματα και από τις δύο πλευρές και το κομμάτι που εντάσσεται στην Επιτροπή την αρμόδια του ΟΣΑ να αναφέρεται σε αυτήν, να κοινοποιείται. Αν πάρουμε 25% του DCI, το μέρος των χρημάτων που αναφέρεται στη σχετική επιτροπή του ΩΣΑ θα ήταν αυξημένο. Και μπορούμε να έχουμε ενισχυμένη συνεργασία. Δεν ξέρω. Ποιος ξέρει. Σε κάθε περίπτωση δέχομαι τη βασική ιδέα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω οι τροπολογίες που υπέβαλα να συμπεριληφθούν. Όμως ανησυχώ μήπως η, Ευρωπα... Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αλλάξει παστικά τον πυρήνα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και σε κατεξαίρεση περιπτώσεις έχουμε περιορισμένη δυνατότητα αξιοποίησης των αναπτυξιακών κονδυλίων για στρατιωτικούς σκοπούς. Αυτή η βασική ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σωστή και πρέπει να τη στηρίξουμε κατά τη γνώμη μου και να προσθέσουμε και κάποια στοιχεία για την αναπτυξιακή χρηματοδότηση και για τις αρχές τις οποίες υπερασπιζόμαστε. Η Πρόεδρος και γι' αυτό ανησυχούσα όταν είδα ότι δεν μας έδωσαν σε εμά την αρμοδιότητα, αλλά την έδωσαν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει επί μακρόν, δεν μπορέσαμε να προοδεύσουμε. Άρα μέσα από τις πολιτικές μας ομάδες πρέπει ο καθένας να δουλέψει για να περάσουμε τις θέσεις μας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Και έχουμε και σύμμαχό μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταληκτική προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η Παρασκευή 5 Μαΐου το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ όλους. Να σας πω ότι αναβάλουμε την εξέταση του σημείου 15 στην ημερήσια διάταξη. Ολοκληρώνεται η συνεδρίαση της Επιτροπής μας και θα τα ξαναπούμε στις 3. Σας ευχαριστώ.